έχω ανακοινώσεις. Πρόταση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά θα προσαρτηθούν στα πρακτικά της παρούσης συνεδριάσεως. Δίνεται τρίμηνη προθεσμία από αύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή από αύριο 21 Ιανουαρίου. Τα πρακτικά της